Λοιπόν, αρχίζουμε γιατί τελειώνει ο χρόνος. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο ε, κατήρτισαν μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής στην Κεντρική Ασία. Θα ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Προεδρία για την ε, πρόθεση που είχε να μάθει τις δικές μας απόψεις πριν εγκρίνει το μήνα αυτό τα συμπεράσματά του το Συμβούλιο η Επιτροπή μας αποφάσισε να συντάξει έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για την Κεντρική Ασία που θα δρομολογηθεί επίσημα τις επόμενες εβδομάδες. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 6 Μαΐου έκανε ακρόαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή, οπότε ε, συμπροματική είναι η σημερινή μας συνεδρίαση. Χωρίς περαιτέρω εισαγωγικά σχόλια, θέλω να δώσω το λόγο στους ε, προσκαλεσμένους μας, τον κύριο Πέλς που είναι ο πρέσβης της Λετωνίας στην Πολιτική Επιτροπή της Ένωσης και στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Δράσης, της ΕΕΒ, τον κύριο Κλάρ. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Κλάρ και στη συνέχεια στον πρέσβη. Δέκα λεπτά έκαστος παρακαλώ κύριε Κλάρ. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι συντομότερος από 10 λεπτά, σας διαβεβαιώ. Because I believe, um, διότι πιστεύω ότι ο κύριος Μπούριαν εκάλυψε το θέμα ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ε, κάλυψε τα όσα και εγώ θα έλεγα για τη στρατηγική αυτή. Ζητώ συγγνώμη προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί ο αρμόδιος διευθυντής για την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία δυστυχώ κολλείεται σήμερα και απουσιάζει, γιατί είναι στη Γεωργία αυτή τη στιγμή και με κάλεσε να τον απληρώσω. Είναι ο Δόκτωρ Βίγκαν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την δυνατότητα που μας δίνετε ε, να είμαστε εδώ σήμερα στα πλαίσια της ολοκλήρωσης αναθεώρησης στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κεντρική Ασία. Είναι μια στρατηγική που το 2007 εγκρίθηκε σε ένα συνολικό έγγραφο για την Ασία και όταν ε, το αναθεωρούσαμε ε, με την πάροδο των ετών εγκρίθηκαν ε, τα αντίστοιχα συμπεράσματα του Συμβουλίου και πιστεύουμε ότι βασικά στοιχεία της στρατηγικής του 2007 τα θεμέλια παραμένουν ακόμα ενισχύει αλλά θα πρέπει να προσαρμόσουμε την στρατηγική ε, στην κατάσταση και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου οφείλουν να το ε, αντανακλούν αυτό. Το βασικό φυσικά ε, ζήτημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η αλλαγή του γεωπολιτικού πλαισίου. Η κρίση στην Ουκρανία και η συγκρουσιακή θέση της Ρωσίας ε, και η ατζέντα που έχουν με την Ευρωσιατική Ένωση οι Ρώσοι να συμπεριλάβουν τις χώρες αυτές, τις κόλπους τους, ε, αφορούν όλες τις χώρες Κεντρικής Ασίας και είναι καιροί δύσκολη και χαλεπή. Ταυτόχρονα όλες οι χώρες αυτές έχουν με διαφορετικό τρόπο και διαφορετικό στυλ ε, ένα πολυπαραγοντικό είδος εξωτερικής πολιτικής από πολλές παραμέτρους. Μέσα σε όλα αυτά εντάσσεται και η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία ήδη έχουν κατατεθεί από την πανεπιστημιακή κοινότητα, think tanks, από την κοινωνία των πολιτών και από τους ίδιους ε, τους εταίρους μας της Κεντρικής Ασίας προτάσεις για την αναθεώρηση. Και το Καζαχστάν και το Ουσμπεκιστάν μας έχουν στείλει αρκετά εκτενή έγγραφα, μάκρος και λέστατα, με τις απόψεις τους για τη στρατηγική σχετικά με την Κεντρική Ασία. Ασία. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το Συμβούλιο συνεργάζονται αυτό το καιρό και ε, προετοιμάζουν το κείμενο των συμπερασμάτων. Αναδύεται ένα έγγραφο που δεν σημαίνει πλήρη ανατροπή ε, του 2007, ε, αλλά γίνεται μια ουσιαστική πολιτική αναθεώρηση του ίδιου εγγράφου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο ρεαλιστικό αλλά συγκεκριμένο ως ε, ε, αναφορά και εταίρος για τη διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι παλιός εταίρος ε, των χωρών αυτών η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει θετική εικόνα. Ιδιαίτερα με, μέσω της ατζέντα μας, της διαφανούς ατζέντα για συνεργασία. φέρω ένα παράδειγμα εδώ. Την περασμένη εβδομάδα συνεδριάσαμε με την, ε, τον, τους επικεφαλής του Ισλαμικού κόμματος του Τατζικιστάν που δεν βγήκε στις εκλογές βουλευτής, δεν κατάφερε να εκλεγεί, αλλά είπε ότι δεν ήταν δημοκρατικές εκλογές και συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, e και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ιδιαίτερη αξιοπιστία, ένα ειδικό βάρος στο Τατζικιστάν και στην Κεντρική Ασία που στερούνται άλλοι παράγοντες όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία, ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι εμάς δεν μας εκλαμβάνουν ως κάποιους που έχουμε ε, σκοπιμότητες ότι θέλουμε κάτι να πάρουμε από αυτούς. Ε, Αλλά ε, ε, είμαστε ειλικρινείς και θέλουμε ειλικρινά και γνήσια να τους βοηθήσουμε. Μπορεί λοιπόν τώρα να αναθεωρήσει η Ένωση τι μπορεί να κάνει ε, συνολικά με την περιφέρεια αυτή ως Κεντρική Ασία και τι μεμονωμένα αναχώρα. Υπάρχουν διαφορές και αυξάνονται αυτές μεταξύ των πέντε κρατών και κοινωνικο-οικονομική τους ανάπτυξη αλλά και η φιλοδοξία που έχουν να συνεργαστούν με την Ευρώπη διαφέρει. Ενισχυμένη συνεργασία λοιπόν και συμφωνία έχουμε με το Καζαχστάν που είναι ένα επίπεδο συνεργασίας ε, στο οποίο δεν έχουμε φτάσει με άλλες χώρες της Κεντρικής Ασίας. Και αυτό είναι επόμενο και φυσικό. Υπάρχουν χώρες που θέλουν πιο στενές σχέσεις και άλλες που θέλουν πιο χαλαρούς δεσμούς. Ε, ε, δεν μπορούμε να έχουμε μια πολιτική για όλους ενιαία, ένα μέγεθος. Ταυτόχρονα Όπως ήδη είπατε, ε, θα πρέπει να συνεχιστούν οι διάφορες πλατφόρμες και τα ε, μέσα που έχουμε περισσότερη ευελιξία, ιδιαίτερα για εκεί που ε, χρειάζονται συγκεκριμένες προσπάθειες. Πάντα με βάση τις ανάγκες και τη ζήτηση από πλευράς τους. Έχει αυξηθεί σημαντικά και η χρηματοδότηση σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 56%. Πάνω από ένα δις είναι για την περίοδο 2014-2020. Η υγιής και αποτελεσματική λοιπόν εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων είναι εκ των όνου κάνευ για να συνεχίσει να έχει επιτυχία αυτή η στρατηγική. Εδώ θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία για την ασφάλεια και τη σταθερότητα συμπεριλαμβανόμένη της αηφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων. Ε, αναφέρθηκε αυτό από το ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η κατάσταση είναι δύσκολη που αντιμετωπίζουν κάποιες χώρες και οικονομικές δυσκολίες αλλά και άλλες. Επιστρέφουν οι μετανάστες από τη Ρωσία. Όλα αυτά πρέπει να τα παρατηρήσουμε πολύ προσεκτικά. Όπως ακούστηκε προηγουμένως, η προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ζήτημα εκεί. Παρά το γεγονός ότι είναι ο πρώτος δωρητής και καμιά φορά και ο πρώτος εμπορικός εταίρος. Πριν από την Κίνα ή τη Ρωσία. Αλλά δεν πολύ φαινόμαστε. Δεν έχουμε αρκετή αναγνώριση για τις ε, προσπάθειες που κάνουμε και αυτό είναι κρίμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να το εξετάσει και να το αντιμετωπίσει όχι μόνο σε αυτή την περιοχή του κόσμου και αλλού. Οπότε και ο διορισμός του ειδικού απεσταλμένου. Ε, και η συχνή του παρουσία στην περιοχή θα βοηθήσει για να γίνει γνωστή περισσότερο και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση και ο χαρακτήρας της και η συμμετοχή της στις χώρες αυτές. Τέλος, το θέμα του συντονισμού και των συνεργειών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των θεσμών δηλαδή με τα κράτη-μέλη και στο εσωτερικό τους και με άλλες χώρες και οργανισμούς και αυτή είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Όπως είπε ο ειδικό ε, απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεργαζόμαστε με τις ε, άλλες διεθνείς οργανώσεις και τους γειτονές τους, με το Συμβούλιο της Ευρώπης, Διεθνή Τράπεζα, τον ΟΑΣΕ, την ε, Ρωσία, Κίνα, Τουρκία και στο μέλλον το Ιράν και το Αφγανιστάν. Θα είναι εξίσου σημαντική. και θα πρέπει αυτό να ε, επιδιωχθεί με έναν τρόπο πολύ καλά συντονισμένο για να επιτύχει η στρατηγική για την Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κλάρ. Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Πέλς. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι της Επιτροπής Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, Ήδη ακούσατε τον ε, πεσταλμένο Μουριάν και γι' αυτό θα περιοριστώ στις απόψεις, στα πράγματα όπως τα βλέπει η Λετωνική Προεδρία. Πρώτον, εκτιμώ ιδιαίτερα την πρωτοβουλία αυτή της Επιτροπής σας να τονιστεί η σχέση μας με την περιοχή αυτή που δεν γίνεται και τόσο συχνά γνωστή. Είναι περιοχή στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ασφάλιση της ασφαλείας και της σταθερότητας, για την προώθηση επιχειρηματικότητας, εμπορίου, καθώς και για περισσότερους δεσμούς με την Ευρώπη, άρα με νέες δυνατότητες πολιτιστικών ανταλλαγών. Γι' αυτό τον λόγο η Κεντρική Ασία θα έπρεπε να τύχει περισσότερης προσοχής και στήριξης από εμά. Η Κεντρική Ασία έχει επιλεγεί ως μία από τις προτεραιότητες της Λετωνικής Προεδρίας. Η ιστορική δεσμή της Λετωνίας με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας the είναι ένα από τα εργαλεία που διαθέτουμε για να προωθήσουμε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την αρχή της Προεδρία εδώ στις Βρυξέλλες η Λετωνία οργάνωσε μία διάσκεψη για την Κεντρική Ασία όπου τονίστηκε η θέλησή μας να ενισχύσουμε τη συνεργασία με την Κεντρική Ασία και να δημιουργήσουμε πιο ανοιχτή και περισσότερη συζήτηση για το μέλλον των σχέσεών μας. Επίσης, η Προεδρία τώρα έφτασε στην τελική της φάση και είναι καλό να γίνει ένας πρώτος απολογισμός. Πρώτον, η ασφάλεια. Ως περιοχή κοντά στο Αφγανιστάν η Κεντρική Ασία έχει στρατηγική σημασία για τη σταθερότητα και την ασφάλεια όλης της περιοχής και γι' αυτό είναι σημαντικό να συνεργαστούμε με τις χώρες Κεντρικής Ασίας για να βελτιώσουμε τη διαχείριση των συνόρων και την ασφάλεια, να καταπολεμήσουμε τη λαθρεμπορία ναρκωτικών και τις τρομοκρατικές δραστηριότητες. Αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Λετωνία θέλησε να παίξει ηγετικό ρόλο στην ομάδα χωρών της Ένωσης για τα επόμενα τρία χρόνια. Αναμένουμε το σχετικό πρόγραμμα να αρχίσει σε δύο εβδομάδες και θα βοηθήσει τις χώρες της Κεντρικής Ασίας να δυναμώσουν τις δυνατότητές τους ελέγχου των συνόρων και σε συνεργασία με την ΙΑΙΕΣ και την Κομισιόν η Προεδρία οργάνωσε σεμινάριο στις Βρυξέλλες για την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών απειλών με εμπειρογνώμονες και από τις χώρες Κεντρικής Ασίας και μετά διοργανώθηκαν συζητήσει στα επίπεδα του διαλόγου υψηλού επίπεδου που έγινε στην Τουσαμπέ. Αναγνωρίσαμε λοιπόν και τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος με την εισαγωγή και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων αντιμετώπισης των κλιματολογικών αλλαγών, το Green Bridge Forum. Η διάσκεψη αυτή μίλησε για την ενδυνάμωση της διαχείρισης του περιβάλλοντος, προστασίας του περιβάλλοντος και της ενίσχυσης δραστηριοτήτων πρασίνης ανάπτυξης. Η γεωργία και η ανάπτυξη της υπαίθρου θεωρούνται προτεραιότητες από πολλές χώρες της Κεντρικής Ασίας για τις σχέσεις τους με την Ένωση. Η γεωργία παραμένει σημαντικό στοιχείο των οικονομιών τους και βασικό έσοδο για πολλούς ανθρώπους στην Κεντρική Ασία. Γι' αυτό η Λετωνία θέλησε να γίνει ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και να χορηγηθούν οι κατάλληλε συμβουλέ. Όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρε Κεντρική Ασία στα θέματα τη καλή διακυβέρνηση και καταπολέμησης της διαφθοράς. Επομένως, κατά την Προεδρία μα οργανώσαμε ορισμένα σεμινάρια σε στενή συνεργασία με τι αρμόδιε οργανώσει από την Κεντρική Ασία. Πριν από λίγε εβδομάδε στη Ρήγα συζητήσαμε θέματα βελτίωσης της διοίκησης των χωρών της Κεντρικής Ασίας όπου ακούστηκαν πολλοί νομικοί εμπειρογνώμονες για να γίνει ανταλλαγή απόψεων και εμπειρίας. Τώρα θα ήθελα να σας τονίσω τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της εδίας. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που έχουν τα ενωσιακά προγράμματα ανώτερης εκπαίδευσης καθώς και επαγγελματικής εκπαίδευσης για την ενίσχυση της ανάπτυξης εκεί κατά τη Λετωνία. Το πρόγραμμα Erasmus Συν είναι, έχει πολλές δυνατότητες και θα μπορούσε να βοηθήσει τις χώρες Κεντρικής Ασίας να ωφεληθούν. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι μαζί με τις υπηρεσίες της Κομισιόν θα οργανωθεί πρόσφατα η πρώτη συνεδρίαση Υπουργών Παιδείας και με την Κεντρική Ασία στη Ρήγα. Αναμένεται η υπουργική αυτή διάσκεψη να δώσει περαιτέρω όθηση και ορμή στη συνεργασία και να αναλυφθούν κοινά προγράμματα για την περίοδο 15 με 17. Το ενδιαφέρον της Λετωνίας για περισσότερη συνεργασία για την παιδεία βασίζεται στην ύπαρξη στενών δεσμών για ανταλλαγές φοιτητών. 925 φοιτητές από την Κεντρική Ασία έχουν γραφτεί σε λετονικά πανεπιστήμια και καλέγια τα τελευταία χρόνια και χάρη στη χρηματοδότηση από τη Λετωνία και άλλες χώρες υπάρχει ειδικό πρόγραμμα και υποτροφίες για της χώρες της Κεντρικής Ασίας και της γειτονίας αυτής. Η βελτίωση των υποδομών μεταφορών είναι τομέας όπου η Λετωνία βλέπει μεγάλες δυνατότητες για συνεργασία με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Οργανώσαμε μια υψηλού επίπεδου διάσκεψη για τις ε, οδικές συνδέσεις μεταξύ χωρών μας και Κεντρικής Ασίας και κατά την Προεδρία θέλουμε επίσης <clears throat> να ενισχύσουμε τους δεσμούς μεταξύ ε, επιχειρηματικών τομέων της Ένωσης με αντίστοιχους της Κεντρικής Ασίας. Η 117η διάσκεψη των εμπορικών επιμελητηρίων έγινε, θα γίνει στις 5 Ιουνίου στη Γιούρμουλα, μια παρεθεριστική πόλη. Και τώρα θα ήθελα να πω μερικά λόγια για την ε, διαδικασία αναθεώρησης των σχέσεων ε, Ένωσης ε, και Κεντρικής Ασίας από την εθνική μας έποψη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί τα τελευταίους μήνες πολλές χώρες μέλη της Ένωσης έχουν εκφράσει ιδέες και προτάσεις και οι χώρες της Κεντρικής Ασίας επίσης. Πολλά ευρωπαϊκά think tanks έχουν επίσης υποβάλει προτάσεις και η Προεδρία επίσης εξετίμησε ιδιαίτερα την πρώτη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής και Οικονομικής Επιτροπής και τη διμερή συζήτηση που θα κάνει η Επιτροπή αυτή ναι, και τώρα για να καταλήξω. Ο κύριοι στόχοι και προτεραιότητες της περίοδου αυτής για την Κεντρική Ασία, η προηγούμενης περίοδου, ισχύουν ακόμη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ανάγκες των μεμονωμένων ε, τη κάθε χώρα της Κεντρικής Ασίας, γιατί δεν είναι όλες δεν έχουν όλες τα ίδια προβλήματα ούτε κοινωνικά, ούτε οικονομικά, ούτε ετοιμότητα ως προς την ετοιμότητα συνεργασίας με την Ένωση. Επίσης πρέπει να διαχωρίσουμε τις διμερείς με τις περιφερειακές συμφωνίες για να έχουμε πιο συγκεκριμένα και αποτελέσματα. Οι πρωτοβουλίε στα τρία θέματα που σας είχα αναφέρει πρέπει να συνεχιστούν αλλά με πιο ευέλικτο τρόπο. Η Προεδρία χαιρετίζει τον οριορισμό του νέου ειδικού εντεταλμένου για την Κεντρική Ασία και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί ήδη προσεκλήθηκε μίλησε στην, ΑΦΕ, στην ΕΠΕΞ. Τέλος, είμαι πεπισμένος ότι μετά την έγκριση των προσεχών συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την στρατηγική της Κεντρικής Ασίας τον Ιουνιό, οι προσπάθειες της Ένωσης για να βελτιωθεί περαιτέρω η εταιρική σχέση με την περιφέρεια της Κεντρικής Ασίας θα αυξηθεί. Η Λετωνία θα συνεχίσει την εμπλοκή της στις χώρες της Κεντρικής Ασίας και μετά την Προεδρία διασφαλίζοντας έτσι ότι όλες οι πρωτοβουλίες και τα σχέδια που άρχισαν υπό εκείνη θα συνεχιστούν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μέσσερς έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε για τόσο πλήρη και αισιόδοξη θα έλεγα παρουσίαση που μας κάνατε. Ε, χαίρομαι που έχουμε αυτή τη συζήτηση. Θα υπάρξει έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για αυτό το θέμα και τυχαίνει να είμαι εγώ εισηγητής. Δεν είναι περιοχή μεγάλης προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ξέρουμε όλοι. Είναι όμως μια περιοχή προτεραιότητας και εξαρτάται και από τις πολιτικές μας για άλλες περιοχές η αναθεώρηση του 2007 είχε τονίσει τα θέματα ασφάλειας Αφγανιστάν. Αυτή τη φορά φαντάζομαι ότι θα ασχοληθούμε περισσότερο με τη σχέση με τη Ρωσία. Τέσσερα πράγματα θέλω να σημειώσω. Πρώτον, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου να συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις περιφερειακές και διμερείς μας σχέσεις εκεί στην περιοχή. Γιατί είναι μια περιοχή που αντιμετωπίζει πάρα πολλές προκλήσεις αυτού του τύπου. Κάποιες υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, κάτι αλλάζει, για κάποιες άλλες δεν αλλάζει τίποτα. Το Καζακστάν ίσως είναι μια μικρή εξαίρεση, ακόμα και εκεί θα έλεγα μεσαία. Δεύτερον, πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία στην αναθεώρηση της στρατηγικής μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, ανάμεσα στην περιφερειακή και τη διμερή προσέγγιση. Γιατί δεν μπορούν να γίνουν όλα καλύτερα σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά ούτε και όλα μπορούν να γίνουν καλύτερα σε διμερές επίπεδο. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν η σωστή ισορροπία στην προσέγγιση αυτή. Πολύ σημαντική δουλειά. Να δούμε δηλαδή πού μπορούμε να έχουμε ευέλικτα πλαίσια εφαρμογής. Τρίτο θέμα. Χρειάζεται περισσότερη συμμετοχή των χωρών μελών. Γιατί δεν είναι μεγάλη προτεραιότητά μας. Γιατί οι χώρες μέλη έχουν ελάχιστες σχέσεις με την περιοχή. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό δεν είναι πολύ ενθαρρυντικό. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά κρίμα. Τα τελευταία 8 χρόνια καμία χώρα μέλος δεν θέλησε να παίξει ηγετικό ρόλο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Και η Λετωνία είναι πολύ καλό που θέλει να κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Και είμαι κι εγώ αισιόδοξο για την προτεραιότητα που βάζει η Λετωνία. Πάντως όντως αυτή είναι μια επένδυση με την οποία μπορούμε να επηρεάσουμε και απέναντι στη Ρωσία και απέναντι ε, στους υπόλοιπους στην περιοχή. Τέλος, όπως είπε και ο πρέσβης Μπουριάν, η αύξηση του μέσου ανάπτυξης και συνεργασίας πάνω από ένα δισεκατομμύριο για την επόμενη περίοδο είναι κάτι σημαντικό. Αλλά πρέπει να προσέξουμε πού θα πάνε τα χρήματα αυτά. 40 ε, δισεκατομμύρια έχει δώσει η Κίνα. Πώς θα ανταγωνιστούμε ένα τέτοιο ποσό. Άρα το δικό μας το ποσό πρέπει να φροντίσουμε να το δαπανίσουμε με αποτελεσματικό τρόπο. Και δεν ξέρω γιατί έχουμε τομεακή προσέγγιση στον προπολογισμό, ενώ οι περισσότεροι διεθνείς δωρητές δεν ακολουθούν την ίδια διαδικασία στην περιοχή. Μα έχει τόση ενδυμική διαφθορά η περιοχή. Δεν είναι κάτι που φέρει καλά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία που μου δώσατε και ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας. Ο κύριος Πέτερ λέει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πρόεδρε θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου πρώτα απ' όλα προς την Λετωνική Προεδρία. Και αυτό γιατί δείχνει μεγάλη προσοχή προς την Κεντρική Ασία. Και συμφωνώ και εγώ με τον κύριο Μέσεριτς για το ότι είναι μία από τις προτεραιότητές μας. Δεν είναι αν μη τι άλλο επειδή είναι γειτονικέ μας χώρες. Συμφωνώ επίσης και με τον κύριο Κλάρ για το πόσο μεγάλη σημασία έχει το κράτος δικαίου. Και πολύ χάρηκα πριν που άκουσα τον κύριο Μπέρντ να αναφέρεται σε ε, καταχώρα αντιμετώπιση. και σε αυτήν την περιοχή η χρηστή διακυβέρνηση πρέπει να είναι ένα όρο κλειδί. Είναι και δικιά μου γνώμη ότι σε μια χώρα όπως το Κυργιστάν που έχει δείξει αρκετά ισχυρές δημοκρατικές φιλοδοξίες και όχι μόνο πρόσφατα θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε περισσότερο στην ανάπτυξη με πιο στοχευμένες δράσεις. Φοβάμαι ότι χάνουμε τη μάχη για την Κεντρική Ασία. Και είμαι και εγώ υπέρ ε, της αντιμετώπισης κατά περίπτωση. Όχι μόνο γιατί οι χώρες αυτές δεν θέλουν να τις βάζουμε στο ίδιο καλάθι όλες, ούτε καν να ονομάζονται όλες μαζί Κεντρική Ασία. Τι νομίζετε λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω για να στηρίξουμε το Κυρκιστάν, το οποίο είχε συγκρούσεις δύο φορές όπως ξέρετε. Δεύτερον, πιστεύετε ότι στο Ουσμπεκιστάν το θέμα της παιδικής εργασίας εξακολουθεί να είναι τόσο σημαντικό. Είχα την εντύπωση ότι είχε υπάρξει κάποια πρόοδος. Και ότι θα έπρεπε να ξαναδούμε την άποψη που έχουμε επ' αυτού για αυτή τη χώρα. Αν υπάρχει πρόοδος δηλαδή ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε ο κύριος Μαμικίνς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, στα λετωνικά. Θέλω να ευχαριστήσω. Ε, θέλω να ρωτήσω κάτι τον εκπρόσωπο της Λετωνικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ για την ε, παρουσίασή σας και την έκθεσή σας. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όταν άρχισε η Λετωνική Προεδρία βάλαμε στο ίδιο τσουβάλι ε, δύο μεγάλες προτεραιότητες, την Ανατολική Γειτονία και την Κεντρική Ασία. Και τώρα μετά από πέντε μήνες έγινε η Σύνοδος Κορυφής για την Ανατολική Γειτονία στη Ρήγα, πραγματικά υψηλωτά του επίπεδου. Από, τη μια. από την άλλη η κεντρική Ασία ήταν λίγο σε δεύτερη μοίρα. Ήταν σε χαμηλότερο επίπεδο οι συσκέψεις και οι συνομιλίες. Γιατί αυτό. Μήπως απέτυχαν οι πρωτοβουλίες μας. Γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δούμε αποτελέσματα. Για την παιδεία και το πρόγραμμα έρασμος. Εντάξει, καλά πάνε, κάπως καλύτερα τα πράγματα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, να σας φάω το χρόνο, αλλά θα μπορούσατε να μας πείτε τι θα μπορέσετε να κάνετε τώρα στην τελική ευθεία, στο τελευταίο μήνα της Προεδρίας, για να αναβαθμιστεί όσο γίνεται αυτή η υπόθεση Κεντρικής Ασίας. Κύριο κύριος Μπίχνερ, σας ευχαριστώ πολύ ε, πολύ ενδιαφέρουσε η έκθεση σας, η παρουσιάση σας. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρκετά προβεβλημένη και ορατή εκεί στις χώρες. Και θέλω να ρωτήσω για δύο συγκεκριμένα μέτρα. Το πρώτο αφορά τη Γερμανία στην περίοδο αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι Αμερικανοί ε, αποκεντρωμένα ε, ήρθαν και ίδρυσαν ε, κάποιες, και ανέλαβαν κάποιες πρωτοβουλίες και είχαν πολύ καλή επαφή με τον τόπιο πληθυσμό, εκδηλώσεις, διοργάνων κτλ. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα σε αυτές τις χώρες. Δεύτερο, έχουμε πολύ θετικές εμπειρίες με ασκούμενους από το Αζερβαϊτζάν. Ε, οι χώρες αυτές έχουν πολύ καλό δυναμικό, πολύ καλά μυαλά, μορφωμένους ανθρώπους και μπορούν να έρθουν να ε, διδαχθούν από μας, να δουν πώς ε, δουλεύουμε. Και όταν γυρίσουν πίσω όμως αυτοί είναι αγκάθη στη σάρκα των κυβερνήσεών τους κάθε φορά που δεν είναι και τόσο φορουμένοι από δημοκρατικές αξίες και ιδεώδη. Ε, τι γίνεται λοιπόν με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την παρουσία ανθρώπων από τις χώρες αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Για να απαντήσετε λοιπόν θα σας ξαναδώσω το λόγο. Έχετε πέντε λεπτά με την αντίστροφη σειρά. Ε, πρώτος ο κύριος Πέλτς. Well, uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Με την άδεια του Πρόεδρου να σας δώσω και κάποια στοιχεία για να απαντήσει και ο κύριος Κλάρ. But regarding the questions, uh, first... Ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συμφωνεί απολύτως η Προεδρία ότι ο διάλογος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθεί ε, σε όλες τις ε, επαφές που έχουμε με τους συνομιλητέ μας από την Κεντρική Ασία και σε πολυμερέ και σε διμερέ επίπεδο. Το κλειδί της επιτυχίας ενδεχομένω είναι αυτό. Να παραμένουμε πάντα σταθεροί, να εκπέμπουμε το ίδιο μήνυμα ανεξαρτήτως συνομιλητού και ε, ομολόγου κάθε φορά, σε διάφορα επίπεδα και με διάφορους τρόπους. Μετά. για την εκπαίδευση και άλλες τομεακές πολιτικές. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για τη Λετωνική Προεδρία για θέματα παιδείας. Ποιο είναι εδώ το κλειδί για να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Είναι ακριβώς αυτή η τομεακή προσέγγιση. Δεν μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ υψηλού επίπεδου μεγαλόστομες πολιτικές δηλώσεις, αλλά η καθημερινή δουλειά στην πράξη σε τομεακές ε, πολιτικές και η συμμετοχή των κρατών μελών ε, με συγκεκριμένη βοήθεια τι συγκεκριμένες δραστηριότητες σε αυτούς τους τομείς. Είναι κρισιμοτάτη. Και ελπίζουμε και η πλατφόρμα αυτή για την παιδεία να ε, επιταχυνθεί τώρα ε, στο εξή, και, άλλωστε για το λόγο αυτό την υιοθετήσαμε και εμείς κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Σε ό,τι αφορά την ε, χρηστή διακυβέρνηση και τις κυβερνήσεις, συμφωνώ απολύτως. Πώς θα μπορούσα άλλωστε να διαφωνήσω. Είναι βασικό στοιχείο που μπορεί να συνεισφέρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ιδιαίτερα για το Κυργιστάν. Πρέπει να αναρωτηθούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε η Κυργιζία αλλιώς. Διότι από τη μια έχει πολύ καλές επιδόσεις ε, στην πορεία προς πιο δημοκρατική εκπροσώπηση στην κοινωνία. Βέβαια από την άλλη, πώς να το πω, εμφανίζει κάποια αστάθεια. Και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποστηριχθούν και ε, να βοηθηθούν οι δομές. Τώρα, τι άλλο με ρωτήσατε. η ε, ανατολική γειτονία και η εταιρική σχέση σε σχέση απέναντι με την Κεντρική Ασία. Είχαμε όντως πρόσφατα τακτικές συνόδους κορυφής για την ανατολική εταιρική σχέση και λιγότερο για την Κεντρική Ασία. Δεν μπορώ όμως να συμφωνήσω με το επιχείρημα που λέγει ότι δεν ήταν σε αρκετά υψηλό επίπεδο οι επαφές. Γιατί στη Ρήγα είχαμε συνεδρίες Υπουργού Μεταφορών με τις χώρες Κεντρικής Ασίας. Και τέλη Ιουνίου, σε υπουργικό επίπεδο και πάλι θα γίνει Συμβούλιο Υπουργών ε, Παιδείας με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Η δική μας προσέγγιση ποια είναι λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η τομεακή δουλειά, η επιμέρους και όχι τα θεωρητικά και τα μεγάλα λόγια. Και όταν αυτό δεν μπορεί να γίνει σε περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να γίνεται διμερός. Σε την οποιαδήποτε σύνθεση. Το θέμα είναι έχουμε συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα. Μου θυμίζουν ότι και οι Υπουργοί Περιβάλλοντος ε, ε, ήρθαν στη Ρήγα μετά από πρωτοβουλία του Green Bridge Forum. Αυτά νομίζω καλύπτουν τις περισσότερες ερωτήσεις σας. Κοίτα, uh, uh, το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι ευγνωμονούμε τα κράτη-μέλη για τις προσπάθειές τους και Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, στρατηγική. Δεν ήταν τόσο αυτονόητο αυτό ότι θα συνέβαινε. Πάντως χαιρόμαστε για τις εξελίξεις. Κατά τη διάρκεια του δικού μας εξαμήνου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Πέλς. Πέντε λεπτά και ο κύριος Κλάκη να απαντήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα επαναλάβω απλώ ότι το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ζωτικό πράγμα και φυσικά αναπόσπαστο τμήμα κάθε μας προγράμματος προς τις χώρες αυτές η καλή διακυβέρνηση επίσης αναφέρθηκε και αυτή είναι τονίζεται στις προτάσεις που υποβάλλουμε στα κράτη-μέλη και χαίρομαι γιατί ανταποκρίθηκαν και ενδυναμώθηκαν μάλιστα. Mm. Η καλή διακυβέρνηση είναι ζωτική, το ξαναλέω, για την ανάπτυξη των χωρών αυτών. Όχι για μας, όχι για μας, για να μπορέσουν εκείνοι να ελκύσουν επενδύσεις, γιατί αλλιώς, αλλιώς λέγω, δεν θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο που να ελκύει Ευρωπαίους επενδυτές. Και η καλή διακυβέρνηση φυσικά είναι από τα θεμέλια για τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι πράγματι πολύ καλό που η Λετωνική Προεδρία προώθησε αυτό το θέμα με την υπουργική διάσκεψη και επίσης ωφελεί, θα είναι χρήσιμο και η Πολωνία που είπε ότι είναι διατεθειμένη να παίξει ηγετικό ρόλο για το εκπαιδευτικό. Μέχρι τώρα κανένα κράτος μέλος δεν είχε αναλάβει τέτοια πρωτοβουλία και είναι πολύ σημαντικό οι Κινέζοι που χορηγούν 40 δις, ναι, φυσικά είναι πολύ ενεργοί στην Κεντρική Ασία, γιατί είναι στη γειτονία τους. Αλλά αυτά τα ποσά να μην τα πιστεύουμε πλήρως, διότι η εξωτερική βοήθεια της Ένωσης δεν είναι μόνο το ένα δις που ανέφερα πριν και τα κράτη-μέλη διμερώς δίνουν λεφτά θα έλεγα ότι κακώς υπολογίσαμε τους αριθμούς προηγουμένως, δεν τονίσαμε δηλαδή παρά μόνο ότι δίνουμε συλλογικά. Έπειτα οι Κινέζοι, τα κινέζικα ποσά συμπεριλαμβάνουν και δάνεια. Αν θέλουμε λοιπόν να προσθέσουμε και τα δάνεια που δίνουμε από τα διάφορα χρηματοπιστωτικά μας ιδρύματα, καταλήγαμε σε ακόμα ψηλότερους αριθμούς. Α μην έρθουμε σε ανταγωνισμό τώρα με τους Κινέζους για αυτά. Έχουμε διαφορετικό πρόγραμμα, η Ένωση έχει διαφορετικό ρόλο και αναγνωρίζουμε ότι ο ρόλος αυτός είναι διαφορετικός και χαιρόμαστε γιατί εμεί δεν έχουμε πολιτικό πρόγραμμα όπως οι άλλοι γείτονες των κεντροασιατών. Στην Κυργίζια υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Είναι η μόνη χώρα που ε, έκανε εκλογές που θεωρήθηκαν ελεύθερες και δίκαιες. Αλλά βέβαια τώρα υπάρχει το νομοσχέδιο για τους ξένους και αυτό μας ανησυχεί και το θέσαμε στους Κυργιζίους το θέτουμε πολύ συχνά και θα συνεχίσουμε να το θέτουμε. Δεν είναι θετικό αυτό. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι η χώρα αυτή θα παραμείνει θα παραμείνει λέγω στο σωστό δρόμο. Ναι. Αλλά βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε εμεί τη δουλειά τους, στη θέση τους, εκείνοι. Εκείνοι εμείς να τους υποστηρίξουμε μπορούμε για την παιδική εργασία στο Ουσβεκιστάν πράγματι τα ακούσαμε αυτά και με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και την Παγκόσμια Τράπεζα θελήσαμε να απαλληθεί η παιδική εργασία στο Αφγανιστάν, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας με έλεγχο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για την καλλιέργεια βάμβακος και όπως είπα και εμεί και η Παγκόσμια <coughs> Τράπεζα ασχολήθηκαν και αυτό είναι καλό. Τέλος. Um, Όσο για το Αμέρικα Χόιζερ, στην Αρμενία υπήρχε ένα τέτοιο πρόγραμμα και φυσικά είναι κάτι που μπορούμε να το εξετάσουμε. Η ορατότητα είναι πρόβλημα για μας και όπως σας είπα όχι μόνο για την κεντρική, στην Κεντρική Ασία αλλά και σε πολλά μέρη του κόσμου. Πρέπει και αυτό να το δούμε και ίσως να είναι σωστός τρόπος αυτός. Ευχαριστούμε πολύ τους προσκεκλημένους μας. Έτσι ολοκληρώνεται η συνεδρίασή μας. Θέλω να σας πω πότε θα συνεδριάσουμε και πάλι. Έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση στις 11 Ιουνίου στο Στρασβούργο, όπου θα ψηφίσουμε διάφορες εκθέσεις και στις Βρυξέλλες συνεδριάζουμε και πάλι 15 και 16 Ιουνίου και 22 και 23 Ιουνίου. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ και ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος.